και είπαμε ότι θα, κάποιες επιτροπές επίσης έχουν ζητήσει ε, διαπραγματεύσεις δύο οργανικές με το 69 γάμο παραγραφός 1 και ε, όλα αυτά υπάρχουν, εντολές δηλαδή, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και θα γίνει και η σχετική καταχώρηση στα πρακτικά της Συνόδου. Σύμφωνα με το άρθρο 69 2 του κανονισμού ενό περισσότερων πολιτικών ομάδων ε, βουλευτέ, όταν φτάσουν στο κατώτερο προβλούμενο όριο, μπορούν να ζητήσουν ε, έγγραφα μέχρι ε, το μεσάνυχτα της 6ης Φεβρουαρίου την ψηφοφορία της αποφάσεως να ξεκινήσουμε τις εν λόγω διαπραγματεύσεις. αν δεν ζητηθεί ψηφοφορία, τότε οι επιτροπές μπορούν να αρχίσουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, σας ενημερώνω ότι την Τετάρτη πρόκειται να συνυπογράψουν τον πρόεδρο του Συμβουλίου ένα νομοθέτημα σύμφωνα με τη συνήθεια νομοθετική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού μας. Ο, ε, ο, ε, τίτλος του νομοθετήματος θα δημοσιεύει.